president Good morning, colleagues. The sitting is now... Καλημέρα συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα στην μερίσια διάταξη είναι δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άστρο και τη μετανάστευση λαμβανόμενης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Τσιότ, ε, εξ του Συμβουλίου. Έχετε τον λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάσταση μεταναστευτική στη Μεσόγειο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των αφήξεων. Συνολικά το 2018 γύρω στις 150.000 ε, παράτυπες αφήξει καταγράφηκαν στα εξωτερικά μας ε, σύνορα στη Μεσόγειο. Αυτό είναι μια πτώση κατά 25% σε σχέση με το 2017 και είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 5 χρόνια. Το σύνολο αυτό του 2018 ήταν επίσης 92% ε, χαμηλότερο από το ιστορικό ύψιλο του 2015. Αυτό μας δείχνει πως η αποφασιστική μας δράση και εμπλοκή με χώρες εταίρους έχουν αποδώσει καρπούς και πρέπει να συνεχιστούν. Ο αριθμός των θανάτων στην θάλασσα βεβαίως παρά είναι ακόμα υψηλός και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να μειωθεί. Αλλά ο αριθμός αυτός ε, του 2018 έχει επίσης μειωθεί κατά 25% σε σχέση με το 2017 και στην κεντρική μεσογειακή οδό έχουμε μείωση πάνω από 50%. Είπατε αρμοστία το ίδιο για τους πρόσφυγες. Υπολογίζω το 2015 η Λιβιακή ακτοφυλακή διέσωσε 50.000 άτομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως παίζει ένα σημαντικό ρόλο και θα ήθελα να αναφερθώ στις πρόσφατες εξελίξεις ε, που αφορούν την Λιβύη και το καταπίστευμα για την Αφρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει 338 εκατομμύρια ευρώ σε έργα σχετικά με τη μετανάστευση στη Λιβύη. 318 υπό το κατεπήγον κατεπίστευμα για την Αφρική και 20 ως διμερή βοήθεια. Το ένα τρίτο, 91 εκατομμύρια δόθηκαν για να στηριχθεί η ακτοφυλακή της χώρας υπομορφήν εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον εξοπλισμό για να, υπάρξει, να υπάρξουν εγκαταστάσεις στην Τρίπολη και να συσταθεί ένα κέντρο ε, διάσωσης ε, θαλάσσιας. Η επιχείρηση Σόφια έχει εκπαιδεύσει 237 ακτοφυλακές μέχρι στιγμής ε, και η ΕΑΖΟ έχει επίσης ε, κάνει εκπαίδευση για την πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου. Όσον αφορά την Λιβύη, ένα σημαντικό τμήμα του προγράμματος ε, είναι 137 εκατομμύρια ευρώ σε υπηρεσίες βοήθειας, σε αποκλεισμένους μετανάστες επίσης, καλύπτει την εθελοντική επιστροφή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που αφορά και την επανένταξη από την οποία έχουν ωφεληθεί πάνω από 16.000 άτομα το 2018 και πάνω από 19.000 άτομα το 2017. Η στήριξη η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως ε, την ε, εκένωση και μεταφορά των ε, μεταναστών μέσω της υπατσαρμοστίας του ΟΗΕ. Από όταν ξεκίνησε το 2017 έχουν ωφεληθεί μέχρι στιγμής πάνω από 2.800 άτομα. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2018 μετά από μήνες διαπραγματεύσεων η υπατερμοστία του ΟΗΕ πάλι με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπόρεσε να ξεκινήσει μια εγκατάσταση συγκέντρωσης και αναχώρησης στην Τρίπολη. Πρόκειται για το πρώτο ανοιχτό κέντρο στη Λιβύη που φιλοξενεί μετανάστες ε, που αφήνονται ελεύθεροι από τα κέντρα κράτησης ε, εν ώψη της μετακατάστασης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρόλα αυτά παραμένουν αρκετές προκλήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές διόδους και είναι πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη. Το Ευρωπαϊκό Τα συμπεράσματα... Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθορίζουν ξεκάθαρες προτεραιότητες. Άρα θα συνεχιστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών στην ανατολική δίωδο και στην κεντρική, στην ανατολική, κεντρική, στην ανατολική δίωδο οι αριθμοί παραμένουν ε, χαμηλοί. Αν και έχουμε σημαντική αύξηση των παράτυπων αφήξεων στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, κάτι το οποίο δείχνει ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για αλλαγές σε αυτήν την δίωδο το πλαίσιο αυτό η συνεργασία με την ε, Τουρκία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν κέρια σημασία. Η συνεργασία μας με τις γειτονικές μεσογειακές χώρες, τα πιο επίγοντα ζητήματα, έχουν συμπληρωθεί με τις επαφές μας με χώρες ε, παραπέρα στην Αφρική. Ο περιφερειακός ε, διάλογος τα τελευταία χρόνια, οι διαδικασίες του Ραμπάτ και του Χαρτούμ, το σχέδιο δράσης της Βαλέτας, είναι χρήσιμα πλαίσια για μια συνολική συνεργασία με τους Αφρικανούς εταίρους. Συμπληρώνονται από σοβαρή χρηματοδότηση μεταξύ των οποίων ε, και το καταπίστευμα για την Αφρική μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι νέες πρωτοβουλίες ε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται όπως η Υπουργική Διάσκεψη της 21ης-22ης Ιανουαρίου που θα συνεισφέρει τις ε, σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών του κόσμου και επίσης ε, θα δημιουργήσει ένα τακτικό φόρμα για συζητήσεις ε, με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την μεταρρύθμιση των κανόνων ασύλου, το Συμβούλιο έχει εργαστεί εντατικά επί των ε, ζητημάτων αυτών σε διαδοχικές προεδρίες. Έχουν λάβει χώρα διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατέληξαν σε σημαντική προόδο σε πέντε από αυτές τις προτάσεις. Ε, με συγχωρείτε κυρία μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να σέβεστε την ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ε, δεν έχετε τον λόγο. Συνεχίστε. η Ρουμανική Προεδρία είναι έτοιμη να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες για να σημειωθεί πρόοδος όπου αυτό είναι δυνατόν. Για άλλα σημαντικά νομοθετικά ζητήματα όπως ο κώδικας Σέγγεν, ο κώδικας Βίζας, ο κανονισμός περί εξηματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Σκοπεύουμε να συνεχιστεί ο διάλογος με το Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές όσον αφορά την μεταρρυθμίση της Ευρωπαϊκής Φυλακής, ε, οι συνομοθέτες συνεργάζονται για να καταλήξουν σε μια θέση που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις. Όμως υπάρχουν ακόμα ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών σε κάποια σημαντικά ζητήματα, όπως παραδείγματο χάρη οι κανονισμοί του Δουβλίνου. Όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν στην σημασία του να βρούμε την σωστή ισορροπία μεταξύ τη ευθύνη και της αλληλεγγύη. Μέχρι στιγμή δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε έναν συμβιβασμό στα συγκεκριμένα στοιχεία της ισορροπίας αυτής. Λέγεται ότι θα πρέπει οι αυξημένες ευθύνες των κρατών μελών να αντισταθμιστούν με ένα προβλέψιμο σύστημα το οποίο θα μπορεί να ανακουφίσει τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζουν την κρίση. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για το πώς θα βρούμε έναν μηχανισμό κατανομής η μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης φαίνεται από το ότι παρά την σημαντική μείωση των αφήξεων, εξακολουθούμε να έχουμε υψηλό αριθμό αιτήσεων ασύλου, μεγάλο ποσοστό των οποίων υποβάλλονται σε χώρες άλλες εκτός από τις χώρες πρώτης γραμμής. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δευτερογενείς κινήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν καταλήξουμε σε μια διαρθρωτική λύση για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you, madam. Please, Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, συνάδελφοι, λίγο σεβασμό στον ομιλητή που έχει το λόγο. Μην διακόπτετε, θα λάβετε το λόγο αργότερα. Εγώ έχω το μικρόφωνο και το λόγο και αποφασίζω. Ε, προχωρούμε τώρα στον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Έχετε το λόγο. Είναι αρκετά λεπτό το ζήτημα, γι' αυτό ε, ας προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Έχω την αίσθηση ότι ξαναβρεθήκαμε εδώ συζητώντας το, το ίδιο θέμα σε παρόμοιες συνθήκες. Ωστόσο, ενώ έχει αλλάξει γύρω μας το όλο τοπίο και οι παράνομες αθήξεις έχουν μειωθεί ε, δραστικά, έχουμε και διαφορετικές πολιτικές συμπεριφορές που δεν άλλαξαν με το χρόνο. Και έτσι βρισκόμαστε και πάλι εδώ. Καταρχάς, να δηλώσω που ότι είναι καλό να βρεθεί λύση αυτή που βρέθηκε για την, για τον, για την αποβίβαση των λαθρομεταναστών, των ε, μεταναστών μάλλον που έφτασαν στη Μάλτα από τα δύο σκάφη ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά μην αυταπατώμεθα. 49 άτομα βρέθηκαν σε σκάφη στη θάλασσα επί τρει εβδομάδε δεν είναι αυτό που θέλει να ε, προασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η κατάσταση. Και επίσης είναι ντροπή να σκεφτεί κανείς ότι αυτό συνέβη στη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί τις ανθρωπιστικές αξίες και την αλληλεγγύη. Εμείς πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε υπέρ των αξιών αυτών. Όμω, εάν οι αξίε του ανθρωπισμού και η αλληλεγγύη δεν προφυλάσσονται, τότε η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί. Στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή δεν βρισκόμαστε προσπαθειών για να προάγουμε τι προσπάθειε συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτή η αποβίβαση να γίνει εφικτή. Εγώ ίδιο, νυχθημερών, ήμουν σε διαρκή συνεννόηση με αρκετού υπουργού Επίσης, δημοσίως κάλεσα όλα τα κρατη να επιδείξουν περισσότερη αλληλεγγύη. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε ενώ ανθρώπινες ζωές κινδυνεύουν στη θάλασσα. Πρώτον, θέλω να επενέσω τη Μάλτα. Ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη που όμως εξέφρασε την αλληλεγγύη της και σκοπεύω να την επισκεφθώ πολύ, να την επισκεφθώ πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κρατημέλη που φρόντισαν να γίνει αποβίβαση στην Μάλτα. Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, ε, Σλοβενία, Ρουμανία, Ιρλανδία και Ιταλία. Όλες οι χώρες αυτές εξέφρασαν την ευρωπαϊκή τους αλληλεγγύη με τον πλέον εύγλωτο τρόπο. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να επαθείται σε αθόρμητες επιτόπιες λύσεις όταν μιλάμε για αποβίβαση μεταναστών. Εγώ, όπως ξέρετε, πήγα χθε στην Ιταλία. Είχα επικοδομητικές συζητήσεις με τους εκπροσώπους της χώρας, με τον ε, Πρωθυπουργό Κόντε και τον Υπουργό Εσωτερικών Σαλβίνη. Όλοι έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης. Διότι δεν μπορεί μόνο με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση να ε, διαχειριστούμε αυτήν την κρίση. Η κατάσταση σήμερα ήδη αποδεικνύει τι πρέπει να κάνουμε. Οι παράνομες αφήξεις σήμερα έχουν μειωθεί δραστικά σε αριθμό σε σχέση από την με την προηγούμενη τριετία. 80% λιγότερο από πέρσι. Κι όμως οι πολιτικές αντιστάσεις σήμερα και οι διαφωνίες παραμένουν ισχυρές. Δεν Ζούμε πλέον μια μεταναστευτική κρίση, μια κρίση του προσφυγικού, όπω κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τα πράγματα. Παρόλα αυτά, ενώ είμαστε αποφασισμένοι να μειωθούν οι παράνομε αφήξει προς την Ευρώπη, θα πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι κάποιοι μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να έρχονται, ακόμα και αν οι αριθμοί είναι πολύ χαμηλότεροι σήμερα. Δεν πρόκειται για κάτι που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ωστόσο. Όμω η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχό μα εάν οι χώρε αναλάβουν δράση μεμονωμένε, μόνε του. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε προβλέψιμα, βιώσιμα συστήματα που να λειτουργούν. Γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη να διαφυλάξει τις ηθικές και ανθρωπιστικές της αξίες και υποχρεώσεις. Ενώ θα δημιουργήσει ένα σταθερό, βιώσιμο, που να διαρκέσει στο μέλλον σύστημα για το άσυλο. Αυτή είναι η ουσία της κοινή ε, ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου. που να ολοκληρωθεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθούν προσωρινές διευθετήσεις και διαδικασίες. Αυτές που θα επιτρέψουν να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τις χώρες που είναι πλέον εκτεθειμένες ε, στις πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσουμε ένα σύνολο ε, δυνατοτήτων ώστε να λειτουργεί μέχρι ο κανονισμός του Δουβλίνου να μεταρρυθμιστεί και να λειτουργήσει πλήρως. Τα έχω ξαναπεί αυτά τον Δεκέμβριο και θα συνεχίσω να τα επαναλαμβάνω μέχρι να το πετύχουμε. Τώρα είναι η στιγμή να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και των κανόνων του. Τώρα είναι η στιγμή οι, κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, και στο Συμβούλιο και να σταματήσουν να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπολογίζω στην αμέριστη στήριξη του σώματός σας. Και θα ήθελα να κλείσω εδώ τι παρατηρήσει μου, εκφράζοντα την εγκλωμοσύνη μου στο Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια αυτή τη τετραετία. Χάρη στη δική σα υποστήριξη και τη δική σα αφοσίωση στο σκοπό αυτό, πετύχαμε πολλά, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και στο μέλλον. Δυστυχώ ο χρόνο ε, περνάει ει βάρο μα. Θα πρέπει να βιαστούμε, να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και να κάνουμε τη δουλειά μα. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Πριν να δώσω το λόγο στους επικεφαλείς των ομαδών, δεν θα δεκτώ μπλε κάρτες στον πρώτο γύρο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και αρκετοί συνάδελφοι θέλουν το λόγο στο τέλος της συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντίας Δεμέρα για την ομάδα του ΕΛΚ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αν και η κρίση της Μεσογείου οδήγησε στο να επικεντρωθούμε την προσοχή μας σε άμεσες ανάγκες. Επίσης μας έδειξε τα διαφορετικά όρια των εργαλείων της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης της 16 Κομισιών πυρώθησε 7 προτάσεις για τη μεταρρυθμίση του κοινού συστήματος ασύλου και σήμερα υπάρχουν δυνατότητες πολιτικής συμφωνίας σε 5 από αυτές. Όμως τα κοινοτικά θεσμικά όργανα δεν έχουν την απαραίτητη αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή, αν και αποτελούν ε, πρόοδο στη διαχείριση τη μετανάστευση, μεταρρύθμιση του Eurodac, για το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου, η δημιουργία ενό κοινό πλασίου για ε, την επαναγκατάσταση, μπορούν να προχωρήσουν αν υπάρχει πολιτική βούληση. Όμω πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη μεταρρύθμιση του συστήματο του Δουβλίνου. Καθώ δύο έτη μετά Τη παρουσίαση τη πρόταση από την Κομισιόν, οι αποκλίνουσε θέσει των κρατών μελών συνεχίζουν να παρεμποδίζουν να υιοθετήσει το Συμβούλιο εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο η Ένωση μπορεί να ανακουφίσει την κρίση Ε, το ε, Ταμείο για την Αφρική, ή το σχέδιο ε, επενδύσεων για το εξωτερικό της Ένωσης. Επίσης, έχει προβλεπτεί και αύξηση του προϋπολογισμού στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που μπορεί να φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να ξεχνάμε και την υπογραφή του ε, παγκόσμιου ε, συμφώνου για τη μετανάστευση με τον ΟΗΕ. Όμω ε, χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και αλληλεγγύη για να αποφύγουμε άντρε, οι γυναίκε και τα παιδιά που φεύγουν από του πολέμου, την κλιματική αλλαγή και τον τρόμο να πεθαίνουν στη θάλασσα ή να πέφτουν στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων. Η έγκριση των επτά εκθέσεων και ε, μια δέσμευση ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι σε εγωισμού και μειοπικέ πολιτικέ θα ήταν μια καλή λύση. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φαγιόν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατακαιρματισμένη μας πολιτική ασύλου ε, είναι απάνθρωποι απέναντι στους ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από τους πολέμους ε, και τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, είχαμε μια τραγική ιστορία που αναφέρεται 49 άνθρωποι για 19 μέρες παρέμεναν στην Μεσόγειο και κανένα από τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να επιτρέψουν στο τη να μπει στα ύδατά του στα εθνικά του ύδατα και πολλές μέρες το πλοίο παρέμενε στην ανοιχτή θάλασσα. Παρ' όλα αυτά ε, θα ήθελα να χαιρετήσω την απόφαση των κρατών και της Σλοβενίας που αποφάσισε να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Κάθε τέτοια τραγωδία μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε εκείνη απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση. Αλλά πότε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε μια τέτοια κοινή προσέγγιση. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί το σύστημα ασύλου και πρέπει να ξεπεραστούν τα μεμονωμένα συμφέροντα κάποιων κρατών μελών. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ασύλου που θα διαρκέσει στο χρόνο και μια μεταρρύθμιση πέρασε από το δικό μας κοινοβούλιο πριν δύο έτη. Συμφωνώ κύριε Επίτροπε ότι οι ευθύνε τώρα είναι στην πλευρά του Συμβουλίου. Πόσο παρόμοιες, πόσες παρόμοιες τραγωδίες αναρωτιέμαι χρειαζόμαστε πριν να αναλάβουμε τελική δράση. Θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι, να σεβόμαστε τις ευρωπαϊκές αξίες και να δείξουμε αλληλεγγύη και μόνο έτσι θα έχουμε μια κοινή λύση και κοινή απάντηση. Σας ευχαριστώ για μισή λεπτό. Εκ μέρου ε, των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θα δώσω το λόγο στην κυρία Στίβενς. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Βλέπουμε μια επανάληψη. Εδώ πέρα αναφέρομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Φερχόφστατ ε, το προηγούμενο καλοκαίρι ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρυθμισής των ευρωπαϊκών ε, κανόνων ασύλου και μετανάστευσης και τότε κατηγόρησε το Συμβούλιο και την ίδια στιγμή ζήτησε ευρωπαϊκά κέντρα σε αφρικανικές χώρες διέλευσης όπου θα μπορούν οι μετανάστες να ζητούν άσυλο. Ε, πραγματικά έτσι θα, δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα. Παγκοσμίω υπάρχουν 60 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δεν μπορούν να, δεν μπορούν να τους δεχτούμε όλους στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει κάποιο όριο. Αλλά έτσι όπως τα θέλει ο κύριος ε, Φερχόφστατ θα παραμείνουμε με ανοιχτά τα σύνορα και θα περιμένουμε το Συμβούλιο να καταλήξει κάπου. Το Κοινοβούλιο προτείνει κάποιες ηλίθιες και ανεφάρμοστες λύσεις ε, περί αερογέφυρας από την Αφρική στην Ευρώπη πάρα πολλά θέματα έχουν κολλήσει στον τομέα της μετανάστευσης. Είναι η στιγμή για ρεαλισμό. Πρέπει να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη είσοδος. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να φυλάξουμε τα σύνορά μας και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εκ μέρους ε, του Άλντε, η κυρία Βίξτρομ, για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ. Πριν από 1,5 χρόνο αυτό το κοινοβούλιο με μια πλειοψηφία δύο τρίτων ε, ενέκρινε μια πραγματιστική μεταρρυθμίση ε, του κανονισμού του Δουβλίνου μετά από πολύ δύσκολη και σκληρή δουλειά. Πέντε ομάδες συμφώνησαν σε ένα κείμενο που ανέφερε την ανάγκη για πραγματικό ευρωπαϊκό συμβασμό. Εμεί υπερψηφίσαμε μία πρόταση που θα διασφάλιζε την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, όπου κάθε κράτο μελός θα έπαιζε ένα θετικό ρόλο στο να διορθώσει τι αποτυχίε του σημερινού συστήματο. Βελτιώσαμε την πρόταση τη Κομισιόν, διασφαλίζοντα ε, άμεση καταγραφή και έλεγχο ασφαλείας των ετούντων ασυλού και μία εξισορρόπηση, μειώνοντα την πίεση στα κράτη-μέλη πρώτη γραμμή και ίσο επιμερισμό των ευθυνών σε όλου. Το δικό μα κείμενο θα έδινε κίνητρο στου ετούντε άσυλων να συνεργαστούν με τι αρχέ αντί ε, να του οδηγήσουμε στη διαφυγή και να πέφτουν στα χέρια των διακινητών. Αυτό που θέλω να δω είναι ένα έφτακτο σύστημα στην Ευρώπη για το άσυλο και όσοι χρειάζονται προστασία ακριβώς να λαμβάνουν την προστασία αυτή και όσοι δεν ε, συμμορφώνονται με τα κριτήρια, δεν πληρούν τα κριτήρια, να στέλνονται πίσω. Εμείς ε, κάναμε τη δουλειά μας ε, στο Κοινοβούλιο, αλλά τι έκαναν τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά όλο ένα και περισσότερο κατέβηκαν ε, στα χαρακόμματα και όλα φαίνεται να ανησυχούν κυρίως για τον εαυτό τους και κανένα δεν είναι έτοιμο να βρει συμβιβασμό. Τώρα θα παραθέσω τον κύριο Βραμόπουλο. Ανοίξτε τα μάτια σας ε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε χαμηλά ποσοστά μετανάστευσης και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι λίγοι που φτάνουν στις ακτές, στις ακτές μας και πρέπει να τους αναλάβουμε πλήρως και θα πρέπει να το κάνουμε από κοινού. Το αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα από τη δράση των κρατών μελών είναι ότι οι άνθρωποι που διασώζονται στη θάλασσα θα πρέπει να περιμένουν εβδομάδε σε πλήρη κατάσταση απελπισία, καθώ τα κράτη-μέλη τσακώνονται για το μέλλον του και φαίνεται κάθε φορά ο πύχη να τίθεται όλο ένα και χαμηλότερα. Πιστέψτε με, θα έρθει η μέρα τη κρίση και οι μελλοντικέ γενιέ θα μα ρωτήσουν όλου μα γιατί επιτρέψατε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί. Κανένας ε, δεν μπορεί να δώσει μια πλήρη απάντηση σε αυτό. Αλλά ξέρουμε ότι κατορθέσαμε να δημιουργήσουμε συστήματα για τα πάντα εκτός από ε, τους ανθρώπους. Όμως έχει έρθει η μέρα για μας να παρουσιάσουμε αποτελέσματα. Thank you. Ευχαριστούμε. Και τώρα εκ μέρους των Πρασίνων για δύο λεπτά ο κύριος Λάμπερ. Λάμπερ. Ευχαριστώ. Ε, ήταν νύχτα και ε, έπρεπε να ανέβω σε ένα κανό. Ε, έβλεπα πολλούς οι οποίοι προσπαθούσαν να πιαστούν από που μπορούσαν. Άνθρωποι που φώναζαν, ούρλιαζαν, έκλεγαν. Νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Αυτή είναι η μαρτυρία ενός μετανάστη που διασώθηκε στη Μεσόγειο. Όλες τις μέρες στα σύνορα της Ευρώπης μας οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή απλώς ήθελαν να ξεφύγουν από την κόλαση. Ε, περίπου 18.000 από το 2014. Εάν η Ευρώπη δεν μπορεί να ε, υποδεχτεί όλο τον πόνο που υπάρχει στον κόσμο, θα πρέπει να αναλάβει το μερίδιό τη, το μερίδιό τη ευθύνη για να αντιμετωπίσει τα γενεσοργά αιτία τη μετανάστευση. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πρωταθλητή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν διστάζει να γίνει μεγαλύτερη σύμμαχο των ε, καθεστώτων καταπίεση όπω το Σουδάν ή τη Ερυθρέα ή αποτυχημένων κρατών όπω η Λιβύη. Σήμερα με τα ευρωπαϊκά χρήματα χρηματοδοτούμε χώρε με ένοπλε συμμορίε που τι έχουμε βαφτίσει εκτοφυλακέ. Ε, μία ε, απάτη η οποία όμω δεν ξεγελά κανέναν. Ο στόχο μα είναι ξεκάθαρο να εμποδίσουμε την παραμικρή αίτηση για άσυλο προ την Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχο που ξεκάθαρα ανακοίνωσε ο Αυστριακό Υπουργό Εσωτερικών τον περασμένο Ιούλιο. Αλλά α μην αυταπατώμαθα. Αυτό είναι ακροδεξιό και οι σχέσει του έχουν εγκριθεί παρόλα αυτά από τι ε, θέσει των αρχηγών κατών και κυβερνήσεων τη δεξιά και τη αριστερά. Στην Σύνοδο, κυρία Υπουργέ, είδατε ότι η επιτυχία τη πολιτική ασύλου και μετανάστευση ήταν μόνο ε, η μείωση των αφήξεων. Η Ευρώπη χειρό είναι μια προσβολή στι αξίε μα. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ε, θανατηφόρα αυτά καθεστώτα, τα φωνικά καθεστώτα που ποδοπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ε, και να μην του μοιάσουμε. Είναι ήδη ίσω αργά για το Βέλγιο και την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Γαλλία, όπου ορισμένε κυβερνήσει αποδίδουν ευθύνε στου μετανάστε μετανάστε και βοηθούν. Εδώ και ένα χρόνο ο καθένας ε, απορρίπτει ε, με απλοϊκές τοποθετήσεις την αλληλεγγύη, ενώ το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία έχει εγκρίνει την ε, έκφραση της αλληλεγγύης και θέλει να αποφύγει την λαϊκιστική προσέγγιση. Θα πρέπει λοιπόν να εγκαταλείψουμε τους εθνικούς εγωισμούς και να κάνουμε περισσότερα. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα και πρέπει να κάνει περισσότερα. Διότι αυτό το περισσότερο και το καλύτερο επιβάλλεται αν δεν θέλουμε να χάσουμε τις αξίες μας. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Και τώρα για την Γκουε, η κυρία Ένστ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτά τα οποία είπατε, αλλά τι ήρθε σήμερα να μας πει το Συμβούλιο. Έχουν πνιγεί 14.000 άτομα τα τελευταία χρόνια στα εξωτερικά σύνορα. Γι' αυτά έρθετε να μας πείτε. Για τα εξαφανισμένα παιδιά, τα χιλιάδες παιδιά που ε, απλά εξαφανίστηκαν σε αυτές τις επισφαλείς οδούς για τους βιασμούς γυναικών στις λιβικές ε, φυλακές. Θέλετε να μιλήσετε για αυτά τα πράγματα στο Συμβούλιο. Εσείς μπλοκάρετε εδώ και 1,5 χρόνο όλες τις προτάσεις που έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία 2 τρίτων. Και όχι μόνο το Δουβλίνο και την οδηγία εισδοχής. Μπλοκάρετε την προοδευτική πολιτική ασύλου. Είστε συνένοχοι Δρέπομαι για λογαριασμό σας στο Συμβούλιο. Και πραγματικά ε, δεν δικαιούστε να ομιλείτε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Και τώρα για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας για να λεπτό η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου έχει ε, καταπατηθεί από τους, Ευρωπαϊ... από εθνικούς εγωισμούς που δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε κοινές θέσεις για, τον... για την κατανομή των ε, ευθυνών για την έκφραση αλληλεγγύης με την πολιτική ασύλου και μετανάστευση των κατών Αυτό το ορίζει και το άρθρο 80 της συνθήκης άλλωστε. Βάσει πρόσφατης μελέτης της EPRS, η ε, στάση των 100 μελών όχι απλώς τις ανθρωπιστικές αξίες καταπατούν, αλλά έχουν και οικονομικό κόστος, 49 δις ευρώ. Ε, αυτό συμπεριλαμβάνει το κόστος της έλλειψης αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις επανακαταστάσεις του Δουβλίνου, τους επαναπατρισμούς και τις αφήξεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εμποδίσουμε την δράση των εμπόρων ανθρώπων όσων θέλουν να δραπετεύσουν από πολέμους και ε, συγκρούσεις και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να περάσουν από, τις πράξεις, από τα λόγια στις πράξεις μάλλον και να φανούν συνεπείς με τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι συνθήκες, να εκφράσουν την ελληνική τους, να υπάρξει συνεργασία και να υπάρξει και συνέπεια δίνοντας ένα τέρμα στις νέο απεικιοκρατικές πολιτικές που συνεχίζουν να, να αποσταθεροποιούν ολόκληρες περιοχές της Αφρικανικής Υπήρου. Ε, για ίδιον όφελο. Εδώ λοιπόν, ω επιβεβαίωσε ο Ιταλό Πρωθυπουργό Κονπέγερη, ε, ε, χθε, συγγνώμη, ορίζοντα το πρόγραμμα τη μετανάστευση ω ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, είναι κάτι που δείχνει ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε τι χώρε μεμονωμένα να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο. Εάν το κάνουμε αυτό, μπορεί να καταρρεύσει ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Χρειάζονται κοινέ προσπάθειε. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριο Δεγράφ για την Ευρώπη των Εθνών και των Ελευθεριών. Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο και η Κομισιόν επιθυμούν την ε, περαιτέρω μετανάστευση. Και λένε ότι καταφέραμε να περιορίσουμε την μετανάστευση. Είναι όμως απλά το αποτέλεσμα της συμφωνίας με την Τουρκία και της διαφθοράς με δισεκατομμύρια. Και απλά είναι το αποτέλεσμα της σκληρής πολιτικής επίσης του Ματέο Σαλβίνη και το Συμβούλιο προτείνει να φτιαχτούν κάποια κέντρα για την επιστροφή παρανόμων μεταναστών, ενώ η κυρία Μέρκελ την προηγούμενη μόλις εβδομάδα αναγνώρισε ότι αυτή την στιγμή δεν λειτουργεί η συμφωνία με την ε, Τουρκία. Δεν έχουμε καταφέρει να στείλουμε ούτε έναν άνθρωπο πίσω. Πρέπει λοιπόν να έρθει η στιγμή των πατριωτών. Όπω ζητάμε εδώ και χρόνια στον Ολλανδία. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα όχι μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των κρατών μελών. Έτσι δεν θα μπορεί κάποιο να έρχεται ελεύθερα από την Γερμανία στην Ολλανδία. Και θα πρέπει επίσης να επιστρέφονται οι άνθρωποι στις αφρικανικές ακτές, κάτι το οποίο δεν κάνει και δεν θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Η μόνη λύση για αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η συνεργασία κυρίαρχων κρατών. Και λέω σε Συμβούλιο και Κομισιόν, σταματήστε να πετάτε λεφτά και ακολουθήστε την πορεία της Ουγγαρίας, Πολωνίας και Ιταλίας. Τώρα για τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Επτήτος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η ευρωπαϊκή ένωση αν και γνώριζε ότι τα κράτη εισόδου ισπανία ιταλία και ελλάδα δεν έχουν τις απαιτούμενες δυνατότητες εντούτοις ανέχθηκε να παραμείνουν επί μακρό χρονικό διάστημα σε αυτά και κυρίως στην ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδων παρανόμων μεταναστών οι οποίοι ζητούν άσυλο. οι άνθρωποι αυτοί όπως γνωρίζετε ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες κυρίως στην ελλάδα και αυτό αποτελεί στίγμα για τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μας. από την άλλη πλευρά τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο η ευρωπαϊκή ένωση προσπαθεί να μας πείσει ότι θα επιλύσει το πρόβλημα με το να προτείνει κάποιες μεταρρυθμίσεις στο θεσμό του ασύλου και κυρίως στην αναχρονιστική ε, συνθήκη του δουβλίνου. όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν θα επιτύχουν και δεν θα επιτύχουν πολύ απλά διότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση κανένα κράτος δεν πρόκειται να τις εφαρμόσει και θα μείνουν γράμμα και κενό περιεχομένου. διότι ποιο κράτος στην πράξη θα είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση ασύλου; Μα το κράτο εισόδου Πώ θα περιοριστεί η μετακίνηση, η δευτερογενή μετακίνηση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των ανθρώπων, μα φυσικά με το να παραμείνουν στο κράτο εισόδου. Έτσι λοιπόν, κυρίω η Ελλάδα θα παραμείνει και θα μετατραπεί σε ένα χώρο μονίμου εγκαταστάσεω λαθρομεταναστών. Α αφήσει λοιπόν τι σπασμωδικέ κινήσει και την υποκρισία η Ευρωπαϊκή Ένωση και α αφήσει τα κράτη να προστατεύσουν τα σύνορά του και να συνεργαστούν μεταξύ του για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι επιμέρους ε, παρεμβάσεις, η κυρία Βόζενμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι ξέρουμε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα αποτελεί την πενταετία που διανύσαμε μια ρογμή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. πρέπει να μιλήσουμε με αλήθειε. η επιτροπή έχει κάνει πολύ σημαντικέ προσπάθειε και εμεί ω κοινοβούλιο πήραμε καθοριστικέ αποφάσει. όμω το γεγονό ότι ιδιαίτερα για την πρόταση του δουβλίνου που ήταν απόλυτα ισορροπημένη μένει ανοιχτό στο συμβούλιο δείχνει τι ευθύνε των κυβερνήσεων συγκεκριμένων κρατών μελών. πρέπει να αποδείξουμε στι επερχόμενε εκλογέ υπάρχει ικανό διάστημα ότι η αλληλεγγύη και η ίση κατανομή ευθυνών είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών διότι αναμφισβήτητα το γεγονός ότι βιώνουμε μια αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση την καθοριστική του ζητήματος αυτού χωρίς ευθύνη επαναλαμβάνω της επιτροπής ή του κοινοβουλίου ρίχνει ε, νερό στο μήλο του λαϊκισμού και το επόμενο στίχημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να αποδείξουμε ότι στην ευρωπαϊκή ένωση η δημοκρατία μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό λαϊκισμό. προέρχομαι από την ελλάδα που ξέρετε όλοι ότι ήταν πρώτη πύλη εισόδου λόγω της γεωγραφικής της θέσεως και οι δραματικές ροές του 2015 ρυθμίστηκαν πολύ σημαντικά αλλά πάντα το πρόβλημα υπάρχει και μπορεί η κυβέρνηση της χώρας μου να είχε προβλήματα στη διαχείριση και στις ελλειπείς υποδομές όμως είναι η πρώτη χώρα το πρώτο κράτος μέρος που έδειξε την αλληλεγγύη στην πράξη. αυτή η αλληλεγγύη είναι και το στίχημα των επόμενων εκλογών είναι το στίχημα του μέλλοντος της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ανακοινώσω ότι επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δεν μπορούμε να δεκτούμε μπλε κάρτα. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Κάρβερ, αλλά θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε στο Κατσδιάι. Για 1,5 λεπτό, κύριε Βαλενσιάνο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, στρέφομαι στη Ρουμανική Προεδρία για να σας πω ότι εσείς έχετε την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσετε να ρίξετε φως σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πιο δύσκολο να τα κάνετε χειρότερα από την Ευστρική Προεδρία, άρα έχετε μια ευκαιρία γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να συνεχίζουμε να συζητάμε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο οι πολίτες της Ευρώπης πρέπει να ξέρουν ότι έχει κάνει τα καθήκοντά του το Κοινοβούλιο, ότι εμείς έχουμε ένα χάρτη πορεία για να επιλύσουμε τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγειο και στην Αφρική ότι έχουμε μία συνταγή για μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου που να είναι ανθρωπιστική ε, αλλά και αξιοπρεπής και είναι πολλά από τα κράτη-μέλη που φρενάρουν τη λύση αυτή. Είναι σημαντικό να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί οι πολίτες μιλούν για το είναι Ευρωπαϊκή στο σύνολό τη. Όμως δεν μιλάμε για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει τη δουλειά του και η Κομισιόν σε, μεγάλο βαθμό κάνει τη δουλειά της. Το Συμβούλιο μπλοκάρει τη λύση. Μιλάμε για το πρόβλημα της Μεσογείου σαν να ήταν ε, ανθρωπιστικό δράμα. Αυτό λέει ο τίτλος μας, όμως αντί γι' αυτό το αντιμετωπίζουμε σαν ένα απλό τεχνικό πρόβλημα και έχουμε 49 ανθρώπους ε, μέσα στις καταιγίδε ε, του χειμώνα γιατί δεν μπορούμε να τους υποδεκτούμε σε κάποιο λιμάνι μας. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπλοκάρουν μία κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου. Αυτό πρέπει να ξέρουν οι πολίτες για να στραφούν στις κυβερνήσεις τους. Γιατί επιμένω, αυτό το κοινοβούλιο που επίσης αποτελείται από 27 διαφορετικά έθνη και πολλές διαφορετικές πολιτικές ομάδες κατόρθωσε να ψηφίσει μια σημαντική συμφωνία που θα έδινε λύση στο δράμα που βιώνουν αυτή τη στιγμή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Εμείς κάναμε τα καθήκοντά μας, είναι η δική σας σειρά ε, για το Συμβούλιο. Θα ήθελα παρακαλώ να σας υπενθυμίσω ότι πιέζει ο χρόνος. Να σεβαστείτε το χρόνο ομιλία σας. Ο κύριος Χαλάχο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από πολλά έτη συζητήσεων και εργασιών, ακόμη δεν είμαστε κοντά σε μία λύση για τη μεταναστευτική κρίση. Ο λόγος είναι ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου δεν ήταν ρεαλιστικές. Η αριστερά και το κεντρό λένε ότι θέλουν λύσεις οι Ευρωπαίοι. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά οι πολίτες δεν θέλουν κακές λύσεις. Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου επικεντρώνεται σε ιδέες όπως η ελληλεγγύη, η διαχείριση και ο επιμερισμός του άχθους. Αυτό που θέλουν όμως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν είναι απλώς μια μετανάστευση διαχειρίσιμη, αλλά λιγότερη μετανάστευση, γιατί η μαζική μετανάστευση από τον τρίτο κόσμο βλάπτει τις κοινωνίες μας. Η μείωση Τη μετανάστευση θα πρέπει να είναι ο κρεγονίο λίθος οποιασδήποτε ευρωπαϊκή λύση. Αυτό ήδη έχει κατανοηθεί. Έχει γίνει κατανοητό σε πολλά κράτη-μέλη. Ελπίζω το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη βούληση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα που θέλουν οι Ευρωπαίοι και χρειάζονται. σα. ευχαριστώ. Και τώρα, για δύο λεπτά η κυρία Ιντβαλτ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι θα λέγαμε αν 2.000 άνθρωποι έβρισκαν το θάνατο προσπαθώντας να περάσουν ε, το συνεργικό τείχος ε, του κυρίου Τραμπ. Δεν θα το θεωρήσω, θεωρούσαμε τεράστια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ, απ' την άλλη, ακούμε την Προεδρία να λέει «Α, έχει βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση. Μειώθηκαν τα νούμερα». Αλλά, κυρία Πρόεδρε, πέρσι πάνω από 2.000 άνθρωποι πέθαναν προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Και ξέρετε, είμαστε πολύ επικριτικοί και καλά ε, κάνουμε απέναντι στο τείχος του Τραμπ, όμως το φρούριο Ευρώπη αποτελεί ακριβώς ισοδύναμο αυτού του τείχους. Και εσείς στο Συμβούλιο χτίζετε το φρούριο Ευρώπη, χτίζετε το τείχος. Απλώς ε, τυχαίνει να έχουμε τη Μεσόγειο ενδιάμεσα. Τώρα, όπως ο Τραμπ και το ανόητο τείχος του, το Συμβούλιο χρησιμοποιεί το φρούριο Ευρώπη για λαϊκιστικούς σκοπούς, για πολιτική συζήτηση και όπως και ο Τραμπ για το τείχος και εσείς δαπανάτε δισεκατομμύρια για το φρούρο Ευρώπη και χρηματοδοτεί τα δίστακτα καθεστώτα ότι είναι τη δέσμη μέτρων που είναι στο τραπέζι και έχει θετηθεί από το Κοινοβούλιο. Και δεν είναι μόνο το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, είναι και οι τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος του Γκτάνσκ δολοφονήθηκε και καλωσόρισε χιλιάδες μετανάστες στην πόλη του. Θα πρέπει να δείτε το παράδειγμα του και να μάθετε από αυτό το παράδειγμα από όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τις εκκλησίες που ζητούν μια ανθρωπινή και αποτελεσματική πολιτική ασύλου. Σταματήστε λοιπόν να παίζετε παιχνίδια και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ισχυρή προσωπική του δέσμευση και για όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για να μια κοινή πολιτική ασύλου. Έχω όμως ένα μικρό αίτημα από εσά να μην καταθέσετε νέε προτάσει στο τραπέζι όπω είναι ένα διατύπωση τη οδηγία για την επιστροφή. Δεν είναι απαραίτητο και είναι μέρο των ανόητων πολιτικών παιχνιδιών του Συμβουλίου. Να κάνετε αυτό που περιμένουν οι πολίτε από εσά και θετήσετε τη δεσμή μέτρων για το άσυλο, γιατί ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Γερμανία μα το έχει αποδείξει. Απλώ κάντε το λοιπόν. Ευχαριστώ. κύριε Λάμπερτ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τους αριθμούς. Αναφέρθηκαν πριν τα 65 εκατομμύρια. Πρόκειται για τον αριθμό εκτοπισμένων ανθρώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι στην ίδια τους τη χώρα. Και βλέπουμε μια αύξηση στον αριθμό προσφύγων. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων, διώξεων και ε, θα ε, είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και ακόμα και οι πατριώτες θα ήθελαν, νομίζω, μια ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αν ανησυχούν τόσο πολύ για τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων. Ανησυχώ όμως για τα όσα συμβαίνουν στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η αναπτυξιακή μας πολιτική προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στον έλεγχο της μετανάστευσης αντί για μείωση της φτώχειας. Και θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο εάν θεωρεί ότι έχουμε την σωστή ισορροπία. Όταν κάνουμε τα στραβά μάτια στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Τουρκία και Λιβύη, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αρκετά για την επανεγκατάσταση που αναφέρατε και όσον αφορά το Δουβλίνο και τις δευτερογενείς κινήσεις, εάν κάνουμε αρκετά για να μην υπάρχουν οι παράγοντες απόθυσης ε, και όπου δεν ασκούν σωστά την πολιτική ασύλου τα κράτη-μέλη, οπότε ο κόσμος πάει σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη για ένα λεπτό. Λέμε διαρκώς ότι η Ένωσή μας έχει βασιστεί στο δίκαιο. Ψεύδος. Με την μετανάστευση δείχνουμε ότι δεν είμαστε Ένωση και παραβιάζουμε το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Οι κανονισμοί στους οποίους εμένει το Συμβούλιο είναι αυτοί της ασφάλειας των συνοριοφυλάκων και των επαναπατρισμών που ε, εξωτερικεύουν, αναθέτουν εξωτερικό στο σύστημα ασύλου. Καμία έκφραση αλληλεγγύης. Όλα έχουν ισοπεδωθεί. Εδώ και μισή χρόνο το Συμβούλιο δεν έχει κάνει αντιπροτάσεις για την τέταρτη εκδοχή του Δουβλίνου. Στα υπόλοιπα θέματα για την επανεγκατάσταση ας πούμε δεν έχουμε αποτέλεσμα εδώ και ένα χρόνο. Να τα αποτελέσματα τσακωμή μεταξύ των κρατών μελών, η διάσωση στη θάλασσα κατηγορείται και η ανθρωπιστική βοήθεια. Δίνεται βοήθεια για να υλοποιηθούν οι κανόνες του τρίτου Δουβλίνου και ε, οι μετανάστες πηγαίνουν πίσω στα γκούρλακ της Λιβύης. Ε, κανένας δεν νοιάζεται για τους νεκρούς. Ε, το Συμβούλιο είναι ένοχο. Ένοχο αμέλειας ανάληψης των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων του. Έχει δίκιο ο Επίτροπος Αβραμόπουλος. Τώρα είναι η ώρα. Now is the time. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκίλη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπέρ είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε σκάφη και λέμβους για να ξεφύγουν από την κόλαση της Λιβύης. Εάν ήταν ακόμα εδώ, δεν είναι ακόμα στην αίθουσα. Αλλά κύριε Λαμπέρ, αυτό συμπεριλαμβάνει και τους μετανάστες που φτάνουν στη Γαλλία για να περάσουν ε, την ε, μάχη Από τι προσπαθούν να ξεφύγουν. Ποια είναι η κόλαση της Λιβύης στη Γαλλία από την οποία δραπετεύουν. Είναι ετούντες άσυλο είναι μετανάστες απλώς και το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα που είναι διφορούμενο. Θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ψευδοάσυλο. Εάν δεν δούμε την πολιτική μετανάστευση, δεν μπορούμε να στραφούμε στο άσυλο. Πρέπει να έχουμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία για να κρίνουμε πώς έρχονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη, ώστε οι τοπικές αρχές να ξέρουν τι θα κάνουν, ε, θα τους δώσουν στέγη, θα τους βρουν δουλειές, θα τους φτιάξουν σχολεία και θα τους διαθέσουν γιατρούς και δασκάλους, διότι αυτή τη στιγμή είναι όλα τζάμπα. Και το μόνο που καταφέρνουμε είναι όσοι έχουν ανοίξει τα σύνορά του, όπω η Γερμανία, να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν και τελικά τους ε, παραπέμπουν σε άλλα κράτη όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία που δεν τους θέλουν. Δεν τους θέλουν γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές. Πώς θα διαχειριστούμε λοιπόν πραγματικά ε, εδώ χρειάζεται μια πραγματική διαχείριση, ανάληψη ευθύνη. Εάν διαχειριστούμε σωστά τα σύνορά μα, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τον αριθμό των ανθρώπων που έρχονται με τρόπο νόμιμο. Οπότε Πώ θα διασφαλίσουμε ότι όσοι πραγματικά χρειάζονται το άσυλο και τη διεθνή προστασία δεν αγνοούνται και ότι δεν έχουμε κόποση μετανάστευση από του ανθρώπου που τα πληρώνουν αυτά μεταξύ των συμπατριωτών μα και των Ευρωπαίων. Δεν πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας προηγουμένως, διότι αν δεν βελτιώσουμε αυτό το επίπεδο δεν βελτιώνουμε τίποτε. Απλώς αλλάζουμε θέσεις στα χαρτιά στην τράπουλα χωρίς να λύνουμε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μποργκέτσιο για ένα λεπτό. Δεν ε, είναι ο χειρό η Ευρώπη. Θα έλεγα ότι ο χειρό έχει γίνει η Ιταλία. Και ο Υπουργό Αλβίνη τουλάχιστον είναι θαραλέος κατάφερε να εφαρμόσει την λαϊκιστική, όπως τη λένε, συνταγή. Δηλαδή να σταματήσει τα σκάφη, να σταματήσει τους ε, εμπόρους ανθρώπων. Αυτό είναι η πραγματική ντροπή. Και αυτό το έχει επιτρέψει η ίδια η Ευρώπη. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ξέχασε να μας πει και να μας θυμίσει τον κατάλογο των ε, ε, 670 μεταναστών πρέπει να επαναγκατασταθούν ε, και είχε αναλάβει να το κάνει αυτό η Ευρώπη. Πήγε στη Ρώμη για να δώσει εγγύηση στην Ιταλική κυβέρνηση. Και εδώ ε, πολλοί εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη του προ τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Α περάσουμε λοιπόν στην έκφραση τη αλληλεγγύη, ε, στην χειροπιαστή έκφραση. Κύριε Αβραμόπουλε, πείτε μα πόσοι από αυτού του μετανάστε που πρέπει να επαναγκατασταθούν βρίσκονται στην Ιταλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναλάβει να τους ε, μεταφέρει. Πού πήγανε. Μόνο υποκριτές βλέπουμε. Η Ιταλία είναι η μόνη που πρέπει να επομιστεί τις ευθύνες και να πληρώσει το τίμημα των λανθασμένων πολιτικών. Να μπλοκάρει τα σκάφη που φτάνουν για να αποβιβάσουν μετανάστες. Να τους εμποδίσει. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Έχει λήξει ο χρόνος σας. Το Ιταλικό κράτος έχει ε, από τις ε, ανώτερες πολιτικές βουλήσεις άλλων. Συνάδελφοι, αυτό είναι ένα από του λόγου γιατί μπορεί να μην υπάρξει δυνατότητα για το κατσδιάι, γιατί όλοι μιλούν παραπάνω από το χρόνο που του έχει δοθεί. Έτσι λοιπόν, παρακαλώ, σεβαστείτε το χρόνο αγόρευση. Για ένα λεπτό, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Γούλ που θα ακολουθήσει το παράδειγμα μου. Ευχαριστώ. Πάντα προσπαθώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολιτική να ελέγξει τους μετανάστες, αλλά ε, θέλει ε, να ακολουθήσει μια εμπορική πολιτική και τελικά έχει γίνει μια υπηρεσία ταξί για τους διακινητές και τις συμμορίες. Αν επιμένει η Ευρωπαϊκή αν βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες ε, ε, οι αιτήσει ασύλου να ε, κατατίθενται εκτός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα διακοπεί καμέσω αυτή η διαδικασία. Τελικά έχουμε καταλήξει στο να στέλνονται οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καταναγκαστική εργασία. Τώρα οι εθνικοί ηγέτες μπορούν να προστατεύσουν τα έθνη από του εαυτού σα, Ο κύριο Κούρ στην Αυστρία, ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο Ματέο Σελβίνη στην Ιταλία. Αυτοί οι δημοκρατικοί ηγέτε έχουν ξαναπάρει τον έλεγχο από του διακινητέ μεταναστών για του πολίτε. Τα σύνορα ανήκουν στα έθνη. Χωρί σύνορα δεν υπάρχουν έθνη. Απλώ ε, δίνουμε το πεδίο στου διακινητέ και στου λαθρέμπορου να δράσουν. Η κυρία Γκάλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Εμείς ε, θα πρέπει να αποφύγουμε να έρθουν ε, χιλιάδες ε, μετανάστες στα σύνορά μας. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν μπορούν να έρχονται παράνομα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εξαρθρώσουμε τα δίκτυα των διακινητών και να προστατεύσουμε και να ελέγξουμε την Μεσόγειο. Ουσιαστικά εδώ ε, μιλάμε για μια επιχείρηση ε, και τελικά έχουμε και τις ΜΚΟ οι οποίες αναλαμβάνουν ε, τους μετανάστες στο τελευταίο στάδιο του ταξιδιού τους. Είναι σαφές ότι κάθε φορά θα έχουμε όλο ένα και μεγαλύτερα κύματα μεταναστών προς την Ευρώπη και τελικά όπως έχουν τα πράγματα θα διαρκέσει δεκαετίες. Το πρόβλημα και η υποχρεωτική κατανομή των μεταναστών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα λύσει το πρόβλημα ούτε η ανθρωπιστική βοήθεια γιατί τελικά έχουμε ένα παράγοντα έλξης. Όλα αυτά αποτελούν παράγοντα έλξης. Και ξέρουν ε, ότι αν φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά θα τους διαμοιράσουν σε διάφορες χώρες. Εδώ μιλάμε για μη διαχείριση μιας κατάστασης, ε, γιατί τελικά αυτή ε, προωθεί την διακίνηση ανθρώπων. Όμως πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή στις χώρες προέλευσης. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στις χώρες καταγωγής τους. Η κυρία Σλάιν για 1,5 λεπτό. Εγώ θα περίμενα να ξεκινήσει το Συμβούλιο την παρέμβασή του ζητώντα συγγνώμη από τα 49 άτομα και από το πλήρωμα των δύο σκαφών ε, καθώς τους κρατήσετε στη θάλασσα για 20 μέρες. Όμως τελικά είδαμε τα όσα λέτε συνήθως ότι έχουν μειωθεί οι ροές Αλλά αν είναι αυτός ο στόχος σα, ποιος ε, είναι ο επόμενος στόχος να πυροβολείτε κατευθείαν τα σκάφη και θα πρέπει ε, να ντρέπονται οι κυβερνήσει Τη της Μάλτας και της Ιταλίας αλλά και άλλε που δεν ε, επέτρεψαν τον ελιμενισμό των σκαφών αυτών και τελικά αντί να προχωρούμε φαίνεται να υπαναχωρούμε. Είχαν δεσμευτεί οι κυβερνήσει ε, για ε, να προβούν στην μετεγκατάσταση όμως τελικά τα τελευταία δύο χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Χρειαζόμαστε διαφορετικές λύσει και μεταρρύθμιση του Δουβλίνου ψηφίστηκε με πλειοψηφία δύο τρίτων εδώ στο Κοινοβούλιο και ε, επιμερίζει τις ευθύνες με ισότιμο τρόπο και υποχρεώνει κάθε κράτος μέλος να ε, δεσμευτεί να αναλάβει τις ευθύνες του ως προς την υποδοχή. Κυβερνήσεις, κάντε τη δουλειά σας και εγκρίνετε αυτή τη μεταρρύθμιση. Διαφορετικά εσείς θα πρέπει να εξηγήσετε στους Ευρωπαίους πολίτες γιατί η αδράνειά σας ε, την οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Και να ρωτήσω τους υποκριτές όπως ε, τον κύριο Μποργκέτσο τι κάνατε με τις ε, μετεγκαταστάσεις αν έχετε απόσχει, αν έχει απόσχει η κυβέρνησή σα ε, από τις αποφάσει. Ευχαριστώ. Περνάμε στην κυρία Γούνιμπερκ τώρα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι, ότι χάρη σε αυτό το μηχανισμό του Δοβλίνου βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Σήμερα μιλάμε για αλληλεγγύη, αλλά τελικά δεν καταλαβαίνουμε σε τι συνίσταται η αλληλεγγύη. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αλληλεγγύη υποχρεωτικά. Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι κούσια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναγκάσει ένα κράτο μέλο να δείξει αλληλεγγύη με διάφορε ποσοστώσει που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στο τάδε ή στο δίνα κράτο μέλο. Ε, και γι' αυτό βλέπουμε αυτό τον κατακαιρματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω αυτό είναι κάτι που δεν μπορέσαμε ποτέ να το καταλάβουμε. Ότι οι λύσει στο μεταναστευτικό θα πρέπει να επικεντρώνονται σε λύσει που είναι βιώσιμε, που δεν επιβάλλονται. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει πραγματική βούληση και να μην περνά από διορθωτικούς μηχανισμούς, αλλά θα πρέπει να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις που να έχουν νόημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Βαλενσιάνο, θέλετε να αναφέρετε ένα σημείο ε, διαδικαστικό. Είναι κάτι πολύ απλό, Πρόεδρε. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ελάχιστη κοινοβουλευτική ευγένεια. Καταρχήν, ο κύριος Μπερκέτσιο ε, μίλησε παραπάνω και κατόπιν προσέβαλε τους υπόλοιπου βουλευτέ. Εσείς έπρεπε να έχετε παρέμβει, γιατί δεν είναι κάτι αποδεκτό αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο. Όντως, Πολλέ φορές ε, εγώ προσπάθησα να παρέμβω και προσπαθώ να εξισορροπήσω μια πολύ έντονη συζήτηση. Σα ευχαριστώ για όσα είπατε. Ο κύριος Ουρτασούν τώρα για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε για την ε, μετανάστευση. Η Ευρώπη ε, σε πάρα πολλά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Καταρχήν αρνείται να έχει μια πολιτική υποδοχή στο προσφύγων και θα ήθελα και εγώ να ζητήσω από την Προεδρία να απεμπλοκάρει τη μεταρρυθμίση του Δουβλίνου. Δεν μπορούμε να περάσουμε ένα λεπτό παραπάνω. Ξέρω ότι προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο, αλλά πιο αργά θα σας παρακαλώ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το ένα λεπτό χωρίς να έχουμε μια ε, πολιτική υποδοχή. Και δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπική στη κρίση. Αυτό που έγινε με το sea και άφησε γυναίκες και παιδιά στη μέση της θάλασσας για μέρες ε, χωρίς ε, να τους επιτρέπει να ελιμενιστούν ε, είναι κάτι ντροπιαστικό. Και έχουμε τώρα και την περίπτωση του Open Arms, ε, το κράβι αυτό, το κρατάνε στο λιμάνι της Βαρκελόνης και ε, τα κράτη θα πρέπει να σεβαστούν ε, τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Να απομπλοκάρετε λοιπόν το Δουβλίνο και να αφήσετε τις ΜΚΟ να εργαστούν αν εσείς δεν θέλετε να το κάνετε. Σας ευχαριστώ. Thank you. One minute, Mr. Benito. Ο κύριος Μπενίτος Ιλουάγα παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι του Συμβουλίου. Αυτό που κάνετε εσείς δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτική μεταναστευτική και ασύλου, αλλά ε, κλείνετε τα σύνορα και κάνετε εξωτερική ανάθεση. Εδώ μιλάμε για δολοφονίες, ε, είτε πνίγονται στη Μεσόγειο, είτε εγκαταλείπονται στην έρημο. Όλα τη σημασία έχει μετανάστευση, αλλά κυρίως είναι φτωχή. Τον προηγούμενο μήνα μια αντιπροσωπεία της ομάδας μου ταξίδεψε στον Ήγηρα για να γνωρίζει αυτό που εσείς αποκαλείτε το εμβληματικό παράδειγμα στην πολιτική ε,